το κείμενο για να βελτιώσουμε την προστασία των δικαιωμάτων αυτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε, Επίτροπε. Ευχαριστούμε την κυρία Γκάλο και τους συναδέλφους. Αύριο ψηφίζουμε στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερίδια διάταξη είναι η έκθεση του Ζωάου Φερέιρο για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Και να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Κύριε Φερέιρα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, την τελευταία χρονιά για πολλούς λόγους είχαμε πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες που μιλούσαν για πυρκαγιές, ε, πλημμύρες, ε, καταστραφές ε, με τεράστιες συνέπειες για τον πληθυσμό και για το έδαφος και αυτό φυσικά δεν ήταν αποκλειστικότητα του τελευταίου έτους. Στα πέντε χρόνια λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 62 αιτήματα χρηματοδότηση από 22 χώρε. Περίπου το 1 τρίτο αφορούσε την κατηγορία των σοβαρών καταστροφών. οι επιπτώσεις για τον πληθυσμό που πλήττεται, για το περιβάλλον και την οικονομία ήταν αξιοσημείωτε, και πολλές φορές ήταν και μόνιμες οι ζημίες που προκλήθηκαν. Ορισμένε φορές ε, χτυπούν ε, αυτούς που έχουν τα λιγότερα μέσα για να προστατευτούν είτε πρόκειται για κράτη είτε πρόκειται για ε, ανθρώπους. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινοτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των καταστραφών και θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών στον τομέα αυτό, κυρίως ε, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται παρέμβαση στα κράτη-μέλη ε, που είναι πιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο και έχουν λιγότερες οικονομικές δυνατότητες να τον αντιμετωπίσουν και μάλιστα τις καταστροφές οι οποίες ε, προκαλούνται από, ανθρώπου. ανθρώπους. Οι ανθρωπογενείς καταστροφές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ορισμένες φορές ενισχύονται και από πολιτικές οι οποίες ε, δεν ε, επιτρέπουν την καλύτερη δράση μεταξύ ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικές οριζόντιες και στην ε, κοινή αγροτική ε, οι οποίες ε, δεν θα δημιουργούν προβλήματα όπως το παρελθόν. Μέχρι πρόσφατα οδηγούσαν και στην ε, απερίμωση των περιοχών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε εκ νέου αυτές τις πολιτικές. Θα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, να υπάρχει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε συνάφεια με το περιβάλλον ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και ένα επιπρόσθετο όφελος για την προάσπιση του εδάφους. Ε, πρόκειται για μια πολύ σημαντική συζήτηση. Η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική σε αρκετέ επιτροπέ. Συζητούσαμε με του σκιώδει συζητητέ και με όσου ε, συνέταξαν γνωμοδοτήσει για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου όσου έδειξαν ενδιαφέρον και ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν, διότι μια συζήτηση, ε, πρόκειται για μια συζήτηση η οποία έγινε ει και μα έκανε όλου κατά τη πλησιότερου. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα χρηματοοικονομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες και θα, ε, τις καταστροφές και θα διαρθρώσει τα μέσα που έχουμε μέχρι ε, στιγμή στη διάθεσή μας και θα πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες να διορθωθούν καταστάσεις οι οποίες ορισμένες φορές οδηγούν στον κίνδυνο. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ένα συντονισμό μεταξύ αυτών των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και να υπάρχει ε, μία κοινή γεωργική πολιτική, να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την ξηρασία και την απερίμωση και να υπάρχει και μία ε, επιστημονική μελέτη για την προστασία των δασών. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εμπειρία που αποκομίσαμε από τι πρόσφατε καταστροφέ και να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό του Ταμείου Παρέμβαση για να μπορούν να γίνονται πιο έγκαιρα οι παρεμβάσει από αυτό το Ταμείο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το θέμα των καταστροφών ε, πολλές φορές αποτέλεσε αντικείμενο ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλές από τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή ήταν παρούσες σε προηγούμενα ψηφίσματα. Αυτό ενισχύει τη σημασία του κειμένου αυτού. Θα πρέπει να το παρακολουθούμε, να υπάρξει και μια συνέχεια και να περάσουμε στην πράξη. ΦΕΦ μέχρι τώρα έχουν γίνει ελάχιστα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ευθύνε για αυτή την καθυστέρηση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, χρησιμοποιήσει αυτή τη μεγάλη υποστήριξη που έχουμε από, την, ε, από το Κοινοβούλιο και φυσικά την υποστήριξη που θα λάβει χωρίς αμφιβολία στο, ε, στην Ολομέλεια και να γνωρίζει ότι αυτά δεν θα πρέπει να παραμείνουν καινογράμμα αλλά να εφαρμοστούν στην πράξη. Έχω πέντε άτομα που ζητούν το λόγο και θα τους δώσω το λόγο κατά σειράν. Η κυρία Πατράου Νέβες πρώτα. Ξαναξεκινώ και λέω ότι πρώτα είναι η κυρία Πατράου Νέβες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική, ιδίω τώρα, διότι οι ανθρωπογενείς ε, καταστροφές είναι όλο και πιο συχνές και από πλευράς περιβαλλοντολογικής και ανθρώπινης είναι σοβαρές οι επιπτώσεις γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά όσον αφορά την πρόληψη. Ήμουν η συγγήτρια για γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Φερέιρα με τον οποίο συνεργαστήκαμε πολύ καλά και υιοθέτησε πολλές από τις τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας. Μιλάμε τον, για τις επιπτώσεις των ε, ε, θεμάτων αυτών και πρέπει να πούμε ότι ιδίω στη Μαδέρα η Πορτογαλία επλήγει και οι ζημίες ανήλθαν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ε, πυρκαγιές δρασών κόστισαν 350 εκατομμύρια ευρώ. Δεν χρειάζονται λοιπόν μόνο μέτρα πρόληψης όπως αναφέρεται στην έκθεση αλλά κάποιο δημόσιο σύστημα αλληλασφαλίσεως και ένα πιο ευέλικτο ε, ταμείο ε, ελεγγύης. Ο κύριος Λούραν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον συγητή για την έκθεση του διότι ε, είδαμε μία αύξηση του αριθμού και της εκτάσεως των ε, φυσικών καταστροφών εφέτος το καλοκαίρι και οι καταστροφές αυτές προκάλεσαν πολλές ζημιές σε πολλά κρατημέλη και επηρέασαν την υποδη... την την υποδομή, την γεωργική πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν μία πολιτική συνοχής για να καταποτελεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα ιδίως όσον αφορά την ε, συμβολή ή στην πρόληψη ιδίως στα κράτη όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες για να αντεπεξέλθουν μόνα τους είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε των θεμάτων αυτών με ε, ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ελέγχθη ότι έχουν ε, ε, αυξηθεί εκθετικά οι ε, ανθρωπογενείς καταστροφές τα τελευταία χρόνια και πέρυσι είχαμε φοβερές πλημμύρες στη χώρα μου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Μπαρνιέ οι οποίοι μας διέθεσαν χρηματοδότηση. Δυστυχώς δεν, δεν έγινε η ίδια επίδειξη αλληλεγγύης στην Ιρλανδία για να αποφύγουμε να ξαναπλημμυρίσουν τα ποτάμια και ε, ε, είμαστε ακόμη εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της πλημμύρας αν ε, υπάρξει αιτία. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επηρεάσει την χώρα μας για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοια προβλήματα στον μέλλον Δηλαδή δεν πρέπει να σας εγκαταλείψουμε. Έκανε ένα λογοπαίδιο ο μιλητής. Ο κύριος Μικολάσιτζης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια ορισμένα κράτη-μέλη επλήγησαν σοβαρά από τις φυσικές καταστροφές που δεν κόστησαν μόνο μεγάλα ποσά αλλά και ανθρώπινες ζωές λόγω αυτών ε, των φυσικών καταστροφών που είναι μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνος του χρειαζόμαστε ε, ένα ταμείο αλληλεγγύης για να μπορέσει να αυξηθεί η ευελιξία ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το ταμείο αυτό αλληλεγγύης θα πρέπει να υπάρχει περιφερειακή ισχυρή πτυχή ε, διότι όπως ξέρετε οι πυρκαγιές των δασών δεν σέβονται την ε, γραμμή διαχωρισμού του κράτους από την περιφέρεια. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ξέρω βέβαια ότι οι ε, προτάσεις μου πρέπει να συμπληρώσουν τους προλαλήσαντες διότι πέραν των οικονομικών προϋποθέσεων που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να επεξένουμε ή στις ε, ζημιές στην Σαξονία που είναι η πατρίδα μου είχαμε πλημμύρες των ποταμών και εκεί χρειάζεται βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών κατά τρόπον ώστε να συντονιστούν τα προληπτικά μέτρα διότι δεν έχει κανένα νόημα στη μία πλευρά του ποταμού να λαμβάνει κανείς μέτρα όταν ε, λίγα χιλιόμετρα πιο πριν δεν υπάρχει καμία πρόληψη. Θα χρειάζεται λοιπόν καλύτερη επικοινωνία διότι φυσικές καταστροφές δεν σταματάνε στα σύνορα και πρέπει να μπορέσουμε από κοινού να τις αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Τέλος, κυρία Παπαδοπούλου. Σε όσα έχουν λεχθεί θα προσθέσω αυτά που έχουμε γράψει στη γνωμάτευση ω εισηγήτρια τη επιτροπή πολιτικών ελευθεριών δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων. η δική μα συμβολή συνίσταται στο γεγονό ότι πέραν από όλα όσα έχουν λεχθεί όσον αφορά συστήματα έγκαιρη προειδοποίηση ταμεία αλληλεγγύη επιχειρησιακή συνεργασία δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονό ότι πρέπει να ακολουθείται η αρχή τη μη διακριτική μεταχείριση όταν πρόκειται για την παροχή βοήθεια. δηλαδή η βοήθεια που δίνεται σε πληγεί περιοχέ πρέπει να χορηγείται με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή το χρώμα το φύλο τη γλώσσα τη θρησκεία τις πολιτικές ή τις άλλες απόψεις την εθνική ή κοινωνική προέλευση την περιουσία την καταγωγή ή άλλο χαρακτηριστικό των αποδεκτών που είναι θύματα από τέτοιες ανθρωπογενείς ή φυσικές ε, καταστροφέ. επίση υπενθυμίζουμε ότι σε καταστάσει καταστροφή και έκτακτη ανάγκη βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τίθενται σε κίνδυνο και πρέπει να προστατεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε επίσης και για την ελληνική λέξη καταστροφή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Σας το λέω εξ ονόματος της Κρυσταλίνα Τζόρτζεβα, της συναδέλφου που δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε το βράδυ ε, για την εκθεσία αυτή τόσο ενδιαφέρουσα τόσο ισορροπημένη που έρχεται εν το χρόνο, όπως είπατε όλοι, αλλά κυρίως ο κύριος Σέσκι προηγουμένως είδαμε τις θεομηνίες, τις καταστροφές να πολλαπλασιάζονται παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη, στο Πακιστάν, στην Αϊτή και ακόμα και στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό έδαφος, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη και το είπατε και εσείς στις παρεμβάσεις Μαδέρα, ε, Πορτογαλία, ο κύριος Ιάρ επίσης στη Σαξονία και δεν ξέχασα το 2002 όταν ήμουν Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής την Θεομηνία τότε που με έκανε να προτείνω την δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ καλά από τη δημιουργία του. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να υπενθυμίσουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε και θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνουμε τις διαδικασίες και να ενισχύουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις ε, καταστροφές, να έχουμε μια πολιτική ε, πρόληψη, διότι η πρόληψη κοστίζει πάντοτε λιγότερο από την επανόρθωση για να μειώσουμε τις τραγικές συνέπειες αυτών ε, των καταστροφών. Θα πρέπει να έχουμε μια πρόσβαση ισορροπημένη για την πρόληψη, την αντιμετώπιση, την απάντηση κύριε Φέρα, έχουμε κοινοτικά μέσα χρηματοοικονομικά για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες της εθνικές για πρόληψη. Ο κύριος Σουάν ανέφερε περιφερειακά ταμεία που μπορούν να στηρίξουν την πρόληψη και το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο ο κύριος Κέλλη υπενθύμησε τη σημασία και μπορώ να σας πω κυρία Παπαδοπούλου ότι η διαχείριση είναι αντικειμενική και μπορούμε πάντοτε να αξιολογήσουμε τους κανόνες ε, των δεσμεύσεων. Αυτό το Ταμείο αλληλεγγύης που γνωρίζω αρκετά καλά υποστηρίζει επίσης τις κατεπίγουσες δράσεις επανορθώσεων ε, και αποζημιώσεων η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων. Εργαζόμαστε με έναν κατάλογο προληπτικών μέτρων που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη για μια χρηματοδότηση κοινοτική και στόχος μας είναι να αυξήσουμε το βαθμό χρησιμοποίησης των κονδυλίων αυτών όπως η κυρία Πατρονερές το ευχήθηκε να επενδύσουμε στην πρόληψη είναι κάτι το απαραίτητο και επιτρέπει να μειωθεί το κόστος της επανόρθωση και της ανοικοδόμησης είσαι. Όπως είπατε κύριε Φερέρα πρέπει να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία για την χαρτογράφηση των κινδύνων. Προσπαθούμε να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για να εμπνευστούμε από τις υφιστάμενες εθνικές πρωτοβουλίες, να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες αυτές πρακτικές για να έχουμε ένα κορμό ευρωπαϊκό για ε, κινδύνους συγκεκριμένους όπως τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τις ακραίες θεομηνίες μέχρι το 2000 2012 θα ενθαρρύνουμε τις χώρες να υιοθετήσουν μέτρα προληπτικά που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές. Έχουμε μια πράσινη βίβλο για την προστασία των δασών και ένα παρατηρητήριο για την ξηρασία. Πάρα πολλές δράσεις ε, τώρα ε, πραγματοποιούνται για να μετρήσουμε τον αντίκτυπο των καταστροφών και θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά στο μέλλον. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν και ο πρόεδρός της ο οποίος το 2004 μου ζήτησε να εργαστώ για μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής άμυνας, για τσουνάμι, άλλες θεομηνίες και καταστροφές η Επιτροπή με την κυρία Τζόρτζεβα θα παρουσιάσει συντόμως προτάσεις για να ενισχύσουμε την ικανότητα ανταπόκρισης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών και θα εργαστούμε ε, σε προτάσεις για να ενισχύσουμε την πρόληψη. Γι' αυτό αυτό το οποίο θα κάνει η Κομισιό, αυτό που θα προτείνει στα κράτη-μέλη νομίζω ότι ανταποκρίνεται ε, στις ανησυχίες του κυρίου Φερέρα τις ανησυχίες που τονίσατε μετά από όλες τις καταστροφές που γνωρίσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. με τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα για την εισήγησή σας. Θα έχουμε την ψηφοφορία αύριο στις 12. Τώρα έχουμε την τελευταία έκθεση την, και έκθεση της κυρίας Θεοχάρους σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο δρόμος της προόδου.